Καλημέρα, συνάδελφοι. Δεν, έχουν καταφτάσει ακόμη όλοι οι συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά, λέω να ξεκινήσουμε και πρωτού περάσουμε στην ε, ημερήσια διάταξή μας. Θέλω να σας πω κάτι δυσάρεστο. Εύα, βάλε τα ακουστικά σου, παρακαλώ. Εσένα φορά αυτό που θα πω. Είναι δυσάρεστο να αποχαιρετούμε κάποιον από τις γραμμές μας. Η Εύα Σανζουάν, συνεργάτηδα των σοσιαλιστών, μας εγκαταλείπει δυστυχώς. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε επιτυχία, κάθε καλό για το μέλλον σου. Ακούω ότι θα περάσεις στην Ισπανική Αντιπροσωπεία των Σοσιαλιστών. Άρα δεν θα σε χάσουμε και τελείω εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα σε έχουμε όμω εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία. Κρίμα. Παρόλα αυτά όμω σου ευχόμαστε οτιδήποτε, ε, ε, κάθε καλό για το μέλλον σου και έχουμε και μια ανθοδέσμη να σου δώσουμε. Grazie. Thank you, Eva, also for, uh, for us. So, dann können wir jetzt zu unserem... Ωραία. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη μέση σε διάταξη. και σας καλωσορίζω στο εργαστήριο για την προστασία των ανελίκων στην ψηφιακή εποχή που διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Β. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους του τμήματος και ε, εν ώψη της προϊούσας ψηφιοποίησης και της διαθεσιμότητας ψηφιακού περιεχομένου για παιδιά και νέους σε όλο και μικρότερη ηλικία εμφανίζονται νέες προκλήσεις για την προστασία τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε και ένα νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εργαστήριό μας θα ασχοληθεί ακριβώς με αυτά τα θέματα, ε, με πιθανές λύσεις, ε, υπάρχουσες λύσεις ε, και με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτήν την μεγάλη πρόκληση. Έχουμε μαζί μας σήμερα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ήθελα να σας τους ε, παρουσιάσω. Πρώτον, έχουμε μαζί μας τον Brian O'Neill, που είναι Διευθυντής των Υπηρεσιών Έρευνας Επιχειρηματικότητας και Κοινοτομίας του Dublin Institute of Technology, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τον ορισμό της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Έχουμε μαζί μας επίσης Στεφάν Σοντρόν, που ε, είναι ερευνητής στο Κοινό Κέντρο Έρευνας με θέμα ψηφιακή ασφάλιση των πολιτών και θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα της ε, μελέτης με τίτλο «Μικρά παιδιά, ηλικίες 0 έως 8 χρονών και ψηφιακή τεχνολογία». Έχουμε μαζί μας επίσης την Εύα Λίβενς που είναι καθηγήτρια δικαίου και τεχνολογίας στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Γάντης και θα μας ε, παρουσιάσει λύσεις και διλήμματα όσον αφορά την πολιτική της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Και τέλος, Σόνια Λίβινγκστον που είναι καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας στο τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας του London, London School of Economics and Political Science και θα μας παρουσιάσει συστάσεις για την ανάπτυξη λύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων στη ψηφιακή εποχή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρουσιάσεις θα είναι. Κάθε εμπειρογνώμονα θα έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά μετά τις δύο πρώτες ε, παρουσιάσεις, θα κάνουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων και θα πρότεινα να ακολουθήσουμε και πάλι αυτήν την ε, γνωστή διαδικασία ping-pong. Σύντομο ερώτημα, σύντομη απάντηση. Έχουμε διαπιστώσει, το λέγαμε και χτες, ότι η συζήτηση έτσι γίνεται πιο ζωντανή και πιο ενδιαφέρουσα. Θα πρότεινα λοιπόν να το κάνουμε έτσι. Και περνάμε αμέσως στην ε, πρώτη παρουσίασή μας θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, κύριο Ονίλ να μας κάνει την παρουσίασή του και βεβαίως να τηρήσει αν γίνεται και το δεκάλεπτο που του έχουμε αφιερώσει. Καλημέρα. Και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την ε, πρόσκληση. Μεγάλη τιμή που μου επιτρέπετε μαζί με τους συναδέλφους να σας παρουσιάσω τις ε, προτάσεις μας για το σημαντικό αυτό θέμα, στο οποίο έχει δώσει βέβαια προσοχή ιδιαίτερη η Επιτροπή σας. Καθήκον μου σήμερα με την παρουσίαση αυτή είναι να περιγράψω το πρόβλημα της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο και να εντοπίσω κινδύνους ε, και προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στη χρήση του διαδικτύου. Ταυτόχρονα θα ήθελα να αναφερθώ σε μακροπρόθεσμες τάσεις στο κυβερνοέγκλημα το σχετικό με τα παιδιά και το ζήτημα της αντιμετώπισης της πρόκλησης ως προς την ε, ε, ρύθμιση, την νομοθετική και την πλαισίωση αυτού του είδους των εγκλημάτων και γενικότερα τα προβλήματα που μπορεί και που πρέπει ο νομοθέτης και οι αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν. Ξεκινούμε με το αξίωμα ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία, είτε είναι στο διαδίκτυο, είτε είναι διαγραμμική ή μη, με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μπορούν και ε, αξίζει να αξιοποιούν. σε μια κοινωνία που έχει καταστήσει κύριο ορόσημο και προτεραιότητα την ε, τεχνολογία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, έρχομαι να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος ενός σώματος ερευνητών που έχει συνεργαστεί με αρχές αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων στο θέμα αυτό για αρκετό καιρό Έτσι λοιπόν η διαδικασία αυτή της, του εντοπισμού και των ε, πολιτικών επιλογών αλλά και των πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια είναι ένας κύριος στόχος, είναι αυτό το οποίο σημαίνει και, τις και την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση, την υποστήριξη των δεξιοτήτων, την ε, εξασφάλιση μεγαλύτερης αντοχής ούτως υπήν στην χρήση της τεχνολογίας, μετρήσιμες ε, δράσεις που θα συμπεριλαμβάνουν βέβαια και την ομοθεσία που θα αντιμετωπίσει το παράνομο και επιζήμιο περιεχόμενο. Μια διαδικασία λοιπόν σε εξέλιξη. Δύο δεκαετίες εμπειρίας έχουμε μέχρι τώρα συλλέξει. Διαφορετική έμφαση δίνεται αναλόγως της περίστασης από τα κράτη-μέλη, μέτρα προστασίας, μέτρα που είναι σχεδιασμένα για, τον, ε, για τη συγκράτηση και τον περιορισμό του κινδύνου από πιθανώς επικίνδυνες ε, ε, συναντήσεις διαγραμμικές στις οποίες μπορεί να εκτεθούν τα παιδιά μας, αλλά και εξισορρόπηση όλων των μέτρων με το θεμητό δικαίωμα κάθε παιδιού να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία του διαδικτύου. Άρα και προστασία αλλά και υποστήριξη του καλύτερου ίντερνετ. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία κλίμακα του προβλήματος αυτού που χαρακτηρίζεται από την άνευ προηγουμένου δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε μια τεχνολογία καινούρια. Πολλές φορές τα παιδιά είναι πρωτοπόροι σαν γενιά σε σχέση με την χρήση αυτή και ξέρουμε από την παγκόσμια και διεθνή έρευνα που, της οποίας έχει ηγηθεί ο Δόκτωρ Λίβινγκστον ότι τα ποσοστά χρήσεως του ίντερνετ για τα παιδιά ή τους νέους είναι συντριπτικά σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, 71% ή 15-24, έναντι ενό 45 περίπου 100 για τις μεγαλύτερες ε, ηλικίες. Επομένως είναι κεντρικό το θέμα, η χρήση αυτή του ίντερνετ για τη ζωή των παιδιών και αυτό έχει μεγάλη σημασία να το αντιληφθούμε για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα και η διαδικτυακή επικοινωνία έχει πρώτο καθεδρία και επικυριαρχία στην καθημερινή ζωή των παιδιών για την επαφή τους με τους φίλους τους ε, συνομήλικους και την κοινωνικοποίησή τους. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει τελείως ε, την εικόνα σε σχέση με αυτή την ηλικιακή ομάδα, γιατί άλλες ηλικιακές ομάδες δεν παρουσίαζαν αντίστοιχα ε, φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να προσφέρουμε υποστήριξη με βάση δεδομένα, αποδεδειγμένα στοιχεία για την υποστήριξη των παιδιών στην χρήση ενός ε, υλικού που μπορεί να είναι χρήσιμο και για την ανάπτυξή τους, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντάς τα και από τον κίνδυνο που μπορεί να είναι που μπορεί να οδηγήσει σε ζημία το παιδί ή και όχι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητο λέει, ότι θα οδηγήσει σε ε, ζημιογόνο αποτέλεσμα για το παιδί. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος, το risk διακινδύνευση έχει να κάνει με την πιθανολόγηση και όχι με την, ε, την δυνατότητα και όχι την πιθανολόγηση του κινδύνου. Βλέπουμε ότι ο κίνδυνος αυτός, η διακινδύνευση, το risk ε, ενισχύεται όσο περισσότερη επαφή με το διαδικτύο και χρήση του διαδικτύου έχει το παιδί και άρα περισσότερα θέματα έχουν οι αρμόδιοι για τη λήψη των αποφάσεων. Αλλά για να ολοκληρώνω σχετικά σύντομα, μια και δεν έχω περιόριστο χρόνο, σας δίνω εδώ μια ταξινόμηση και κατανομή ανατύπω των διακινδυνεύσεων και ε, της βλάβης που μπορεί να υποστεί ένα παιδί σε πεδίο ευρωπαϊκό έχει γίνει σχετική μελέτη η οποία εντοπίζει περιπτώσεις ή συναντήσεις, επαφές των παιδιών που μπορεί να είναι αποδέκτες και θύματα αλλά ταυτόχρονα και συμμετέχονται σε μία πράξη ε, επιζήμια ή βλαβερή ή όπου μπορεί να βρεθούν σε θέση να προξενήσουν ε, κίνδυνο άθελά ε, τους. Είναι πολύ μεγάλη διακινδύνευση, εκτεταμένη, ποικίλη, αναλόγως διαφόρων περιπτώσεων στους διάφορους αυτούς τομείς. Και εδώ σας δίνω πολύ σύντομα παραδείγματα περιπτώσεων ή προβλημάτων που έχουμε εντοπίσει με μια σειρά από μελετών σε σχέση με κινδύνους που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως προς την εμπειρία που έχουν βιώσει τα παιδιά. επί περιεχόμενο το οποίο καταγγέλλεται από τα παιδιά ως ε, περιεχόμενο που τα έχει φέρει σε δύσκολη θέση, τα έχει κάνει να αισθανθούν άσχημα κτλ. Όχι απαραίτητα μόνο πορνογραφικό. Και εδώ έχουμε ένα, 9, 50% ε, για τα παιδιά 9 έως 16 ετών. Αντίστοιχα η κυβερνοπαρενόχληση, κυβερνο, το, το cyberbullying, κυβερνοεκφοβισμός, που επίσης έχει μεγάλο ποσοστό, αλλά όχι το μεγαλύτερο. Η σεξουαλική παρανόχληση, τα ε, σεξουαλικού χαρακτήρα μηνύματα, έχουν επίσης ε, υψηλό επίπεδο, έχουν μεγάλη συχνότητα. Δυσμενείς συνέπειες για τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Το... Ο κυβερνοεκφοβισμός φαίνεται να έχει επίσης ένα σημαντικό κομμάτι αρνητικής επίδραση στα παιδιά κατά πολλαπλούς τρόπους. Είναι όμως ένα από τα ζητήματα, και είναι ένα από τα ζητήματα που πιο συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Για να αναφερθώ πολύ σύντομα στις εγκληματικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, βλαβερό και παράνομο ή και παράνομο ε, περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να διαχωρίζουμε ανάλογα και με την κλίμακα του προβλήματος, στο κυβερνοέγκλημα λοιπόν που αφορά τα παιδιά. Υπάρχει μία σειρά δραστηριοτήτων στο διαδικτύο που μπορεί να υπάγονται και στον ποινικό κώδικα, όπως επίμονο harassment, όπως διαλογή παιδιών οστιμάτων, θυμάτων, όπως ε, χρήση του διαδικτύου για τη διάδοση εξτρεμιστικής ιδεολογίας. Βεβαίως, κύριο επίκεντρο του, της προσοχής είναι η αντιμετώπιση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκβιασμού παιδιών. Αυτό είναι το θέμα το οποίο απασχολεί περισσότερο τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. και βεβαίως προξενεί πολλές ανησυχίες. Νέο στοιχείο από αξιολόγηση της Europol αλλά και άλλες μελέτες έχει να κάνει με νέους τομείς ε, εγκληματικής δραστηριότητες πέραν, ε, ως μια νέα εκδοχή δηλαδή του των σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος των παιδιών μέσα από το διαδίκτυο είναι αυτό του σεξουαλικού εκβιασμού, δηλαδή είτε με εξαναγκασμό είτε με εξαπάτηση, ε, εξασφάλιση πορνογραφικού υλικού από τα παιδιά, τα οποία μετά, το οποίο μετά χρησιμοποιείται για να εξαναγκαστούν σε ε, σεξουαλικές πράξεις ή δραστηριότητες. Βλέπουμε πολλές φορές να συλλέγεται υλικό και να εντοπίζεται το πιο ευάλωτο και πιο νεαρό σε ηλικία παιδί με πολύ οργανωμένον τρόπο. Και εδώ έχουμε μια από τις μεγάλες προκλήσεις για το νομοθέτη και για τους φορείς τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων στο με αυτό ταυτόχρονα. και εδώ είναι το τελευταίο κομμάτι που έχω στην, περιλάβει στην έκθεσή μου, νέοι κίνδυνοι, προκλήσεις, που εδώ έχουμε να κάνουμε με την παρακολούθηση της τεχνολογίας, με τις νέες προκλήσεις που θα αναδυθούν, ε, τα παιδιά χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία σε όλο και πιο μικρή ηλικία Υπάρχουν νέοι λοιπόν κίνδυνοι για την ασφάλεια, για την, την υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, για τους γονείς, για τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς θα συμμετάσχουν σε αυτά. το ίντερνετ των αντικειμένων, επί παραδείγματι, αποτελεί ένα περιβάλλον νέο, στο οποίο θα πρέπει να γίνει και η επιστημονική έρευνα και να συλλεγεί η εμπειρία εκείνη που θα είναι ικανή ώστε να δώσει καθοδήγηση προς γονείς, προς αρμόδιους λήψη αποφάσεων, προς νομοθέτες η προστασία του ιδιωτικού βίου, η ασφάλεια, η συλλογή δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το περιβάλλον και για να ολοκληρώσω με βάση αυτό τον πρώτο ορισμό του χώρου, του... μάλλον τον ορισμό με βάση τα δεδομένα τα επιστημονικά και την εμπειρία, ε, θα πω ότι έχουμε πολύ λίγες μελέτες σε σχέση με τους νεαρούς, τους πιο μικρούς σε ηλικία χρήστες ε, ή τα κινητά μηχανήματα, φορητά τηλέφωνα του καθεξής, ε, ή εμπειρίες σχετικές με διακινδύνευση και ευκαιρίες. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερες έρευνες, γιατί μόνο πέντε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει εθνικές έρευνες που μπορούν να τους καθοδηγήσουν. Χρειάζονται μελέτες που θα καθοδηγήσουν ε, τις αρχές αρμόδιες για τη λήψη των αποφάσεων σε επιλογές τους. Κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και ιδιαίτερα την έμφαση που δίνεται και την, ε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς ε, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε για την παρουσίαση. Η κυρία Σουτχόν έχει το λόγο. Και πίσω σας που Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις διαφάνειες. Σήμερα λοιπόν όπως ακούσαμε από τον Μπράιαν, η παιδική ηλικία μπαίνει στη ψηφιακή εποχή. Εάν δείτε κάποιες οικογένειες με παιδιά, θα καταλάβετε αμέσως πόσο έχει αλλάξει η εμπειρία τους και τα βιώματά τους λίγα μόλις χρόνια. Άρα είμαστε στα χρόνια της ψηφιακής τεχνολογίας και πολύ μικρά παιδιά μέχρι και μωρά καθημερινά χρησιμοποιούν ταμπλέτες, smartphone ε, και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στη μάθηση, στην ασφάλεια ε, και όλα αυτά, για όλα αυτά έχουν τεθεί πολλά ερωτηματικά. Τώρα, για τους οφήβους και για την προεφηβική ηλικία και τη σχέση τους με το ίντερνετ και το ψηφιακό κόσμο γνωρίζουμε πολλά. Έχουμε κάνει πολλές έρευνες, όμως δεν ξέρουμε τη σχέση με την ψηφιακή εποχή των πολύ μικρών παιδιών. Πώς αναπτύσσουν δεξιότητες, ποια είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζουν, ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν. Για να έχουμε λοιπόν στοιχεία, να γεφυρώσουμε το χάσμα, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013 ξεκίνησε μια μελέτη με τίτλο «Ναι, «Μικρά παιδιά από 0 έως 8 και ψηφιακή τεχνολογία». Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να καταλάβουμε περισσότερο σε βάθος τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τα ψηφιακά μέσα, ποια αντίληψη έχουν τα παιδιά και οι γονείς για το ψηφιακό κόσμο, πώς οι γονείς διαχειρίζονται τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τα παιδιά τους, ποιοι είναι οι συγγενείς και σχετιζόμενοι κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες. Προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μια ποιοτική προσέγγιση με βάση την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις. Για δύο βασικούς λόγους αυτό. Πρώτον, τα παιδιά δυσκολεύονται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και οι γονείς μπορούν να κάνουν έναν απολογισμό μόνο για ένα μέρος της πραγματικότητας που υφίσταται. Οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις είναι το καλύτερο για να καταλάβει κανείς ένα φαινόμενο που αναδύεται και πολύ συχνά παρουσιάζει πτυχές απρόσμενες. Είναι μια μελέτη που εκτάθηκε, επεκτάθηκε σε τρία χρόνια, 14-17, έγινε σε τρεις φάσεις με πάνω από 60 ερευνητές, σε 31 ερευνητικά κέντρα σε 21 χώρες οι ερευνητές δίνουν, ε, κάνουν τη δουλειά τους χωρίς ιδιαίτερη στήριξη από μόνοι τους. Πήραμε συνεντεύξεις από 462 παιδιά 6 και 7 ετών και πιο μικρά αδέρφια και γονέων αυτών, άλλοι 400 περίπου. Και ας δούμε τα βασικά ευρήματα για τα πολύ μικρά παιδιά και την ε, πρώτη παιδική ηλικία. Σε γενικές γραμμές τα μικρά παιδιά έχουν μια ισορροπημένη ζωή και η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνε καταλαμβάνουν μέρος αυτή της ζωής μόνο. Μαθαίνουν πολύ γρήγορα πώς θα αλληλεπιδράσουν με αυτές τις συσκευές, παρατηρώντας τη χρήση των συσκευών που κάνουν τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικοι. Παρόλο που μπορεί να μην γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση και γραφή, αναπτύσσουν τις δικές του στρατηγικές αλληλεπίδρασης, αναγνώριση εικόνα, αναγνώριση φωνή ή οπτική αναγνώριση. Και ουσιαστικά ακολουθούν ένα μονοπάτι δοκιμής και λάθους που εκεί εμπεριέχονται κίνδυνοι και σε αυτή τη διαδρομή μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Υπάρχουν κίνδυνοι αλλά αναπτύσσουν έτσι και δεξιότητες και μάλιστα περισσότερες και καλύτερες από ό,τι οι γονείς. Βλέπουν ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούν την ψηφιακή ε, τεχνολογία τόσο περισσότερα μαθαίνουν και με tutorial, με ψηφιακές διδασκαλικές μεθόδους ε, ε, ε, ενισχύουν την κριτική του σκέψη. Η ψηφιακή τεχνολογία για τα παιδιά είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των άλλων. Video game και βίντεο, YouTube και Google Play. Είναι υπαριθμόν ένα λύση κατά της ανίας, αλλά δεν είναι η μόνη χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για να αποκτήσουν πληροφορίες, όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και για τα ενδιαφέροντά τους, για να τα γεμίσουν, να ε, ε, ικανοποιήσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία τους. Και υπάρχουν ευκαιρίες μάθησης ε, και οι γονείς συμφωνούν μόνο όταν ε, το έχει ζητήσει ρητά το σχολείο, δηλαδή ότι η μέρος των μαθημάτων στο σπίτι είναι να κάνει το παιδί τη συγκεκριμένη ψηφιακή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ορισμένα παιδιά δημιουργούν περιεχόμενο και ενδιαφέρονται να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για να το κάνουν ε, έπρεπε να τους διδαχτεί αυτό και από κάποιον μεγαλύτερο πώς θα δημιουργούν και θα ανεβάζουν περιεχόμενο. Πολύ λίγα παιδιά, η μηνιοψηφία είναι ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ε, τα περισσότερα παιδιά μπαίνουν στα επικοινωνιακά συστήματα της οικογένειας, δηλαδή με την εποπτεία της μητέρας ή του πατέρα μπορεί να δημοσιεύσουν κάτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με το λογαριασμό του γονέα. Ε, έχουν πίεση από, το, από τα άλλα παιδιά και ε, θέλουν και αυτά να μπουν σε συγκεκριμένες διαδικτικές ομάδες. Κάποιοι γονείς συνοδεύουν και πλαισιών τα παιδιά τους σε αυτή τη δράση, Άλλοι όμως δεν γνωρίζουν καθόλου του κινδύνου και αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα να πλοηγούνται και να εξερευνούν ό,τι θέλουν στο διαδίκτυο. Τώρα, από πλευρά γονέων, ε, του ενδιαφέρει η προστασία, περιορίζουν την πρόσβαση και έχουν στήριξη και από κοινού χρήση μαζί με το παιδί. Όλα αυτά σχετίζονται με το χρόνο που διαθέτουν, τη γνώση και τις εμπειρίε τους, αλλά και με το πόσο πολύ είναι αποδεκτή η τεχνολογία στη δική τους οικογένεια ή στην κοινωνία στην οποία ζουν. Οι περισσότεροι γονείς έχουν προστατευτικές στρατηγικές που έχουν να κάνουν με το χρόνο, κυρίως και λιγότερο με το περιεχόμενο. Διότι φοβούνται την αρνητική επίδραση στην όραση, στη συγκέντρωση, στις γνωστικές δεξιότητες, στην κοινωνική συμπεριφορά. Φόβοι που και τα ίδια τα παιδιά εκφράζουν όταν παίρνουν το λόγο. Οι φόβοι των γονέων συνάδουν εν μέρη μόνο με τους πραγματικούς κινδύνους. Μία κατάλληλο περιεχόμενο, δυσκολίες αυτορύθμισης, εκφοβισμός και κυβερνοεκφοβισμός, είναι πράγματα που δεν αναφέρθηκαν ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Οι γονείς που δεν γνωρίζουν τόσο πολλά από ίντερνετ περιορίζουν περισσότερο την πρόσβαση στην τεχνολογία σε σύγκριση με τους άλλους. Αλλά συχνά τα παιδιά ξεπερνούν τα όρια κάθε φορά που τους δίδεται αυτή η ευκαιρία. Ανακαλύπτουν τους, τα password, τους μυστικούς κωδικούς και δεν το λένε στους γονείς ότι τα έχουν ανακαλύψει και τα ξέρουν. Οι ψηφιακώ ενήμεροι γονεί χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία περισσότερο από κοινού με, τους, ε, με τα παιδιά τους, ξέρουν ε, τα ε, σφάλματα, τους κινδύνους, τα θετικά και μπορούν να διαχειριστούν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, τα οποία φαίνεται να αποκτούν πολύ περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες. Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι η ψηφιακή επανάσταση είναι αναπόφευκτη, είναι χρήσιμη, αλλά έχει και προκλήσεις. Ουσιαστικά θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στην εφηβική ηλικία και μάλιστα ε, τότε ίσως είναι πολύ αργά γιατί τα παιδιά εκτίθενται ήδη σε μια πληθώρα κινδύνων πριν φτάσουν στην εφηβική ηλικία. Οι γονείς ξέρουν ότι αυτή η τεχνολογία έχει δυναμικό εκπαίδευσης, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται πλήρως. Όταν τα σχολεία θεωρούν ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα ενεργό εργαλείο εκμάθησης, τότε η κριτική σκέψη και η ψηφιακή ενσυναίσθηση των παιδιών οξύνεται, αλλά τότε και οι γονείς προσφέρουν θετική στήριξη, γιατί το ζήτησε το σχολείο. Και υπάρχουν στο Βορρά οι γονείς ε, που ε, περισσότερο λειτουργούν ως σκαλωσιά προκειμένου το παιδί τους να καταφέρει να οικοδομήσει και να ανέβει ψηλότερα στα σκαλοπάτια και γονεί στο νότο κυρίως που λειτουργούν κυρίως ως φύλακες των θυρών ε, προκειμένου να προστατεύσουν περισσότερο. Ίσως ε, υπάρχει έλλειψη κάποιων ε, δικλείδων, δικλείδων ασφαλείας. Άρα, Σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ άνεση, άνηση και διαφορετική αναλόγως τα παιδιά, τις οικογένειες, τις χώρες και ούτω καθεξής. Είναι πολύ κατακαιρματισμένα και μεταβλητά τα προσόντα τα ψηφιακά των παιδιών. Τα βασικά τα ξέρουν όλοι διότι μιμούνται τη συμπεριφορά των γονέων, ωστόσο Λίγα είναι τα παιδιά τα οποία διδάσκουν ψηφιακές δεξιότητες οι γονείς τους και μπορούν πραγματικά να αποκτήσουν ουσιαστικές ψηφιακές δεξιότητες. Οι τεχνικές και κοινωνικές προκλήσεις ε, δυσκολεύουν την υπεύθυνη λειτουργία στο ψηφιακό κόσμο ε, πρέπει να βελτιώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις διαδώσουμε και μεταξύ των γονιών και των νέων και των διδασκόντων ε, για να ε, καταλαγιαστούν οι ανησυχίες και για να δημιουργηθεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής και της οικογενειακής ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή και περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Η κυρία Σόντροβα, αν μπορεί σε ενα μισή λεπτό θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα αυτό που συζητούμε σήμερα. Γνωρίζουμε ότι τόσο οι διδάσκοντες, δάσκαλοι και καθηγητές, όσο και τα σχολεία εν γέννη, ανησυχούν και προβληματίζονται για το πώς μπορούν και να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να προστατευτούν και τα παιδιά από παρενόχληση ή την κακή χρήση αυτών των τεχνολογιών. Είτε πρόκειται για τον υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά από μια οθόνη, ε, χωρίς να μαθαίνουν τα παιδιά, είτε πρόκειται για την έκθεσή τους ε, σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Νομίζω ότι μία λύση θα ήταν να υπάρξει ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών. Για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες επισκεφτήκαμε την Φιλανδία, όπου μας ενημέρωσαν ε, οι διοργανωτές της επίσκεψης αυτής ότι στην Φιλανδία γίνεται πλέον μια καλύτερη, αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών χωρίς αυτό να σημαίνει ε, ότι έχει επεκταθεί χρονικά ή ποσοτικά η χρήση αυτών των νέων ε, τεχνολογιών. Αλλά δίνεται, εξακολουθεί να δίνεται μεγάλη έμφαση και σε άλλες ε, δραστηριότητες όπως είναι ο αθλητισμός. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, διότι το να βασίζεσαι και να αναθέτεις ε, την επίλυση αυτού του ζητήματος αποκλειστικά και μόνο στους γονείς, προφανώς δεν επαρκεί. Φυσικά και υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, στο πώς προσεγγίζει ο κάθε γονέας το ζήτημα της ε, διαχείρισης των ψηφιακών τεχνολογιών. Άρα από εκεί μόνο μια καταγραφή μπορεί να γίνει, όχι να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για το τι είναι κατάλληλο και τι όχι. Ε, από αυτή την άποψη ε, νομίζω ότι χρειάζεται μια ε, κριτική σκέψη και μια πλαισίωση και καθοδήγηση από τα πάνω των γονέων στο πώς θα χειρίζονται την, τα ζητήματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είναι δύσκολο να εμπλέξουμε τους γονείς, ιδίως όσον αφορά τις τεχνικές αλλαγές, τεχνολογικές αλλαγές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν, δεν είναι νέο φαινόμενο. Το παρακολουθήσαμε και τον 20ο συνέδριο. Νομίζω ότι βασικό στοιχείο είναι το σχολείο. Γιατί αυτό που είδαμε στις μελέτες μας είναι ότι εκεί όπου υπήρχαν παιδιά που παρακολουθούσαν, που επισκέπτονταν σχολεία, όπου υπήρχε μια ισόρροπη σχέση με τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες, εκεί οι γονείς άρχισαν να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία, και τις δυνατότητες που δίνει για τη μάθηση. Και εκεί αφιέρωναν και χρόνο και χρήματα ε, προκειμένου να αξιοποιήσουν ε, υπέρ των παιδιών τους τις δυνατότητες αυτές των ε, ψηφιακών τεχνολογιών. Γιατί πράγματι με σωστή χρήση μπορεί κανείς να μάθει πολλά. Το παιδί αλλά και ο γονέας. Και μπορεί πραγματικά ε, μια τέτοια διαδικασία μέσα με επίκεντρο το σχολείο να οδηγήσει σε ανύψωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι. Συμφωνώ απόλυτα με την συνάδελφο. Οι γονεί, πρέπει και αυτοί να βοηθηθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα να διαδραματίσουν τον ρόλο του ψηφιακού φύλακα και του υποστηρικτή της ανάπτυξης των παιδιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπα και στην παρουσίαση μου, υπάρχει κοινή ευθύνη και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει και ένα δίκτυο αλληλοϊποστήριξης. Τα οι να έχουν ε, στενή ε, και ουσιαστική επαφή και σχέση με το σχολείο προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύονται στη σωστή και την ωφέλιμη χρήση των ε, ψηφιακών τεχνολογιών. Και βεβαίως χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει ανταλλαγή ε, ε, βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου όλες οι πλευρές, όλες οι εμπλικόμενες πλευρές να μαθαίνουν η μία από την άλλη. Ευχαριστώ. Κύριε Σοφρίν. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι σήμερα δίνουμε έμφαση στα πολύ μικρά παιδιά έως 8 ή 10 χρονών. Τι γίνεται όμως με τα, με τα, με τα άλλα παιδιά, τους εφήβους 15-16 χρονών, γιατί νομίζω ότι η πρόσβαση αυτών των παιδιών είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μια 24 ε, ώρη κάποιες φορές ε, ενασχόληση παιδιών με την τεχνολογία. Εγώ όταν πήγαινα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ε, ο μόνος τρόπος για να βρεις τους φίλους σου ήταν να πας έξω στην Αλάνα να παίξεις ποδόσφαιρο. Ενώ και μάλιστα ε, άμα σε καλούσαν και νωρίτερα οι γονείς σου να γυρίσεις στο σπίτι μπορεί και να σε κορόιδευαν οι, οι, οι φίλοι σου. Τώρα όμως πια μέσω των νέων τεχνολογιών ε, τα παιδιά μπορούν να έχουν 24 ώρες το 24 ώρο σχέση με τους ε, συνομιλίκους τους, με τους φίλους τους και αυτό δημιουργεί και προβλήματα. Ε, ε, μπορείτε να μας πείτε ποια από τις δύο ομάδες τελικά των παιδιών έτσι όπως τις χωρίσατε ηλικιακά αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο. Ναι, εμείς επικεντρωθήκαμε στα πολύ μικρά παιδιά γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσεων για το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι όλο και πιο μικρά παιδιά ασχολούνται με το διαδίκτυο ε, και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν τελικά με αυτή την τεχνολογία. Δεδομένου αυτού, η έρευνά μας ασχολήθηκε οι ε, έρευνε μα έχουν ασχοληθεί με την χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους εδώ και 10 χρόνια έχουμε μια πιο ε, σαφή εικόνα για εκείνη την ε, ηλικιακή ομάδα. Ο Μπράιαν όμως ίσως ε, μπορεί να σας πει περισσότερο, γιατί εγώ επικεντρώθηκα στη μελέτη μου σε αυτά τα πολύ μικρά παιδιά, οπότε μας πει καλύτερα ο Μπράιαν. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε περισσότερα και καλύτερα ερευνητικά στοιχεία για τις μεγαλύτερες ηλικιακέ ομάδες. Διαλέξαμε την ηλικιακή ομάδα 9 16 για να ε, μάθουμε πράγματα και για τα τελευταία χρόνια της παιδικής ηλικίας και τα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Έχουμε ένα έγγραφο με τις τάσεις και τις αλλαγές και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους για τους εφήβους. Και έρχεται η έρευνα αυτή να το συμπληρώσει αυτό το έγγραφο, γιατί τις ίδιες εμπειρίες βιώνουν όλο και πιο μικρά παιδιά συνεχώς. Τα ίδια βιώματα, τις ίδιες συναντήσεις έχουν. Και ό,τι συμβαίνει στους μεγαλύτερους είδαμε ότι τελικά έρχεται και σε μικρότερα παιδιά και του συμβαίνει. Και γι' αυτό πρέπει να διευρύνουμε την έρευνα και γι' αυτό άλλωστε το κάναμε. Αυτός ο χάρτης που παρουσίασε ο Στέφαν συμβαδίζει πολύ με αυτά που βρίσκουμε ως ευρήματα για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την προσέγγιση των γονέων, για την γνώση των γονέων, για τα βιώματα των παιδιών ε, σε σχέση με την επαφή τους με την ψηφιακή εποχή και τον ψηφιακό κόσμο. Είναι πολύ μεταβλητή η εικόνα με πολλά και διαφορετικά στοιχεία. Δεν είναι εύκολο να γενικευθεί σε όλη την Ευρώπη και χρειάζεται λεπτομερής ενδελεχής έρευνα σε εθνικό επίπεδο για να φανούν τα, οι διαφορετικές εμπειρίες. Σε γενικές γραμμές πολλά παιδιά έχουν ωφέλη Όμως υπάρχει και μία διαστρεβλωτική εμπειρία σε σχέση με τη μόνιμη χρήση και τη μόνιμη σύνδεση στους εφήβους. Και πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα παιδιά, στην τροτότητα ορισμένων παιδιών. Vielleicht, dass man schon im frühen Kindesalter auch tatsächlich mit Medienkompetenzerziehung. Ναι, Βεβαίω θα πρέπει και σε αυτή την ε, τρυφερή ηλικία να υπάρξει η δυνατότητα να μάθουν ε, μέσα από την βασική εκπαίδευση τα παιδιά να διαχειρίζονται, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν διαφορούς κινδύνους. Κατά τρόπο προσεκτικό. Όχι δηλαδή να δέχονται ότι έρχεται χωρίς να το εξετάζουν. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μαλίνοφ. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω μόνο να αναφέρω κάτι. Ε, γίνεται λόγος για προστασία των ανηλίκων από τους γονείς Χθε. Κάναμε λόγο και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Γιατί είναι πολλές οικογένειες όπου παιδιά, επειδή οι γονείς έχουν φύγει στο εξωτερικό για να, εργάζον, για να εργαστούν, γιατί είναι μονογονεϊκές οικογένειες και πάλι εργάζεται η μητέρα ή ο πατέρα ε, διαρκώς. Πολλά είναι τα παιδιά λοιπόν που μεγαλώνουν με τον παππού ή τη γιαγιά. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τόσο η ηλικία μάλιστα. Ίσως είναι και πιο δύσκολο να δοθεί αυτή η έμφαση στους ε, ηλικιωμένους. Αλλά είναι μεγάλα τα ποσοστά παιδιών που ε, είναι υπό την επιμέλεια των, του παππού ή της γιαγιάς. θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής έχουμε να αντιμετωπίσουμε το παράλογο όσο πιο πολύ όσο περισσότερες δεξιότητες έχουν ε, τα παιδιά, οι γονείς, ε, ο παππούς, η τόσο πιο πολύ είναι και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Υποτίθεται ότι άμα προσφέρουμε δεξιότητες και κριτική σκέψη, αλλά βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Καλή φόρμουλα, αλλά θα ήθελα και απαντήσεις. Όσο περισσότερες δεξιότητες, όσο πιο καλά γνωρίζουν ε, την κατάσταση και, τους, ε, και το, τι περί τους τα περιμένει, τόσο προς τους κινδύνους να λαμβάνουν. Στο ίντερνετ, παραδείγματι. Ένα παράδοξο, ε, ένα οξύμορο το οποίο πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Συνήθω είναι απλά τα πράγματα. Όσο τώρα ξέρει, τόσο καλύτερα, τόσο καλύτερα προφυλάσσεσαι. Περισσότερε δεξιότητε, τόσο καλύτερο. Αλλά εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντω, όντω υπάρχει αυτό το οξύμορο. Μα προβληματίζει. όλους εμάς που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε δουλεύοντας στο πεδίο αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ε, νέους και, τους, ε, και τα παιδιά που χρησιμοποιούν ε, το διαδίκτυο. Ωστόσο δείχνουν τα στοιχεία ότι όσο περισσότερη χρήση, όσο περισσότερε δραστηριότητες, τόσο και αυξάνονται οι κίνδυνοι. Τώρα, ο ίδιος ο κίνδυνος οδηγεί σε βλάβη, αυτό δεν είναι δεδομένο. Και επίσης δεν ισχύει, το ίδιο, δεν, δεν ισχύει η ίδια ε, γραμμική ανάπτυξη σε σχέση με τις δεξιότητες. Γιατί όσο περισσότερες δεξιότητες έχει κανείς, τόσο καλύτερα μπορεί να αντιμετωπίσει και να προλάβει τους κινδύνους. και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι πιο εκτεθειμένα, που είναι πιο τροτά, ε, παρακολουθούν το, τη γραμμή της απόκτησης δεξιοτήτων. Άρα χρειάζεται δεξιότητες, χρειάζεται στρατηγικές ασφάλειας, στρατηγικές ασφάλειας, όλα αυτά στα οποία ε, πρέπει να εστιάζεται η εκπαίδευση. Έχουμε καταγραφές με βάση και την εμπειρία των νέων αλλά και τη δυνατότητα να μάθουν από τους ε, συνομιλικούς τους ε, με πολύ καλά αποτελέσματα παραδείγματι τη μετάδοση γνώσεως, ε, την απόκτηση δεξιοτήτων χάρη στην μετάδοση γνώσεως που έχει επιτρέψει η την προστασία από κυβερνοεγκλήματα κυρία Σοντρό, θα ήθελα να πω ότι μία από τις ε, προκλήσεις είναι ο ρυθμός αλλαγής της τεχνολογίας, εξέλιξης τεχνολογίας και σε αυτό πρέπει να διατηρήσουμε άγρυπνο μάτι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ένα νέο WhatsApp, ένα νέο Facebook μπορεί και αύριο ακόμα να προκύψει, για το οποίο δεν θα έχουμε τα εργαλεία έτοιμα να τα δώσουμε στους γονείς, στα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουν κατά τρόπο ε, ισορροπημένο. Άλλη μια πρόκληση λοιπόν εκεί. Ωστόσο, στρατηγικές, όπως λέει και ο Μπράιν, ε, εκμάθηση από το συνομήλικο ή και παρακολούθηση συνοδείας ε, της τάξης των παιδιών, των γονέων, των δασκόντων για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και χωρίς φίλτρο, αλλά ξέροντας πώς να κινηθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τις γενικές ψηφιακές δεξιότητες τις σχετικές με την ασφάλεια. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Κώστα. Πρέπει να πω ότι πολλοί με απασχόλησαν και αναλογίστηκα τα όσα είπαν και ο κύριος Σονέιλ και η κυρία Σοντρούν ότι έλειπε δηλαδή μία έρευνα που να κάλυπτε τις ηλικίες 0 έως 8, δηλαδή την πρώτη παιδική ηλικία όπως λέμε και τις δυνατότητες για μια ψηφιακή παιδαγωγική ε, μόρφωση, εκπαίδευση. Ε, που ε, λείπει αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί κανείς πλέον να είναι αναλφάβητος ως προς την παραδοσιακή γραφή και ανάγνωση αλλά να είναι γραμματιζούμενος εντό εισαγωγικών πάντα ως προς την ψηφιακή χρήση αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην έχει και την συνείδηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων κυρίως για τις πρώτες αυτές οι παιδικές ηλικίε. Ε, σε αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση. Επίσης είπατε και εσείς και συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην έρευνα γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά στοιχεία. Ε, το άλλο, και βέβαια θα μας πούνε και οι λοιποί ομιλητέ μας, ε, στα διάφορα επίπεδα, είτε είναι το επίπεδο της εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο ή των εργαλείων ε, που καθιστούν πιο υπεύθυνε για τις επιλογές τους τις διάφορες επιχειρήσεις, εταιρείε του κλάδου. και αρχές που μπορεί να εισαχθούν σε διάφορες κοινωνικές πλατφόρμες ε, για να ενισχύσουν την ευθύνη τους εναντί των ανηλίκων και των κινδύνων στους οποίους αυτοί εκτίθενται. Ε, και έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξή. Λέτε ότι μόνο πέντε χώρες έχουν ε, έρευνες, δημοσκοπήσεις για τη χρήση του διαδικτύου από τους ανηλίκους. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε. Ειδικά εργαλεία δεν ξέρω αν υπάρχουν σε άλλες χώρε. Εμείς έχουμε σε επίπεδο εθνικής αρχής ε, μια ειδική επιτροπή που ασχολείται με το διαδίκτυο και τους νέους ε, και άλλα τέτοια μέτρα που μπορούν ε, με αρμόδιες αρχές να δώσουν οδηγίες προς ναυτιλωμένους όπως τα λέγαμε για εκείνους που είναι οι πιο εκτεθειμένοι. Ποια είναι λοιπόν η δυνατότητα να κάνουμε, ποιο είναι ο καλύτερος συνδυασμός, μια καλύτερη προσέγγιση. Προσέγγιση βέβαια προς τον γονέα, προς τον ενήλικα αλλά και άλλες δυνατότητες, κατευθυντήριες γραμμές που μπορούμε να προτείνουμε πέραν του νομοθετικού τμήματος που βεβαίως θα το συζητήσουμε μετά. Κύριε Ονίλ, παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Προσδιορίσατε μια σειρά από στοιχεία που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε ε, μια υποστήριξη πολιτικής υψηλής ποιότητας, υψηλού επίπεδου. Και το Τμήμα Πολιτικής έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά την προώθηση βέλσων πρακτικών, όχι μόνο στο, στο επίπεδο της ε, νομοθεσίας, αλλά και των συστάσεων της καθοδήγησης, κάτι που έχει ωφελήσει ε, πολλούς, πολλές πλευρές στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την συμμετοχή της ερευνητικής ε, κοινότητας μέσω του ορίζοντα 2020 ήταν μια, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Όσον, όσον αφορά τον προσδιορισμό των κοινωνικών προκλήσεων αλλά και των κοινωνικών επιπτώσεων των ραγδαίων καινοτομιών και εξελίξεων στην τεχνολογία. Εδώ πραγματικά ορίζοντας 2020 προσέφερε εξαιρετικές ευκαιρίες ερευνητικά προκειμένου να εξετάσουμε τα ζητήματα που αφορούν στην νεολαία σχετικά με τη χρήση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν και εξασφάλιση ότι και ο κλάδος της ε, οικονομίας θα, της τεχνολογίας δηλαδή θα συμμετέχει ενεργά στον προβληματισμό αυτό. Η βιομηχανία προφανώς και φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης προκειμένου να προσφέρονται σε όλους τους πολίτες αλλά ιδίως στα πολύ μικρά παιδιά και στους νέους ε, αξιόπιστα εργαλεία, ασφαλή ε, εργαλεία, ασφαλές περιεχόμενο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το φαινόμενο αυτό είναι πολυεπίπεδο. Η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι απλώς να εντοπίσουμε συγκεκριμένους κινδύνους στους οποίους θα απαντήσουμε με συγκεκριμένες λύσεις. Χρειάζεται να έχουμε μια συνολική εικόνα και ταυτόχρονα να αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Ε, νομίζω ότι δεν έχω κάτι να προσθέσω εκτός ίσως από το εξή. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την πλαισίωση των νέων εργαλείων για νέους και παιδιά για, και για γονείς. Διότι ο κίνδυνος εδώ είναι ότι αν το εργαλείο που θα τους έχουμε προσφέρει εμείς και που θα αντιαποκρίνεται στις δικές μας προδιαγραφές ενδέχεται να είναι υπερβολικά περιοριστικό. Τι θα κάνουν τα παιδιά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, απλά θα πάνε στην επόμενη πλατφόρμα. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο να το έχουμε κατά νου και να μην το ξεχνάμε. Πρόεδρος, Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Τα μοντέλα κατηγοριοποίησης ε, που χρησιμοποιούμε με βάση την ηλικία ε, αντιμετωπίζουν και έχουν πάντοτε τον κίνδυνο να καθόμαστε και να ε, εξετάζουμε σε αυτές τις έρευνες τους γονείς που ήδη ασχολούνται ή τέλο πάντων προβληματίζονται με αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε τώρα από αυτά που μας είπατε ότι εκείνοι που γνωρίζουν, που, που μάλλον που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν οι ίδιοι τους ψηφιακές δεξιότητες, κυρίως περιορίζουν τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν διάφορες απαγορεύσεις μέσα στο σπίτι ως προς το χρόνο ε, που θα ε, παρακολουθήσουν ή θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες στα παιδιά. Ενώ το αντίθετο, γονείς που ξέρουν και έχουν ψηφιακές δεξιότητε κυρίως συνοδεύουν τα παιδιά τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το κάνουν από κοινού δηλαδή. Μπορείτε δηλαδή με βεβαιότητα να πείτε ότι το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο του γονέα επηρεάζει τη στάση του μέσα στο σπίτι του και τους κανόνες που, θα, που ορίζει για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είναι αλήθες. Και ήταν και ένας από τους στόχους της έρευνας, να δούμε πώς ανταποκρίνονται οι γονείς, πώς ε, ε απαντούν στα αιτήματα των παιδιών. Η πιο ενεργή και υποστηρικτική διαμεσολάβεση εξαρτάται από το κατά πόσο οι γονείς είναι ενημερωμένοι, είναι ψηφιακώς ενήμεροι, αλφαβητισμένοι και όχι αναλφάβητοι ψηφιακά. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για τα διάφορα είδη γονέων και τις γνώσεις τους. Και ε, ρωτήσαμε τα παιδιά κατά πόσο νιώθουν ότι ξέρουν ακριβώς τόσα όσα ξέρουν οι γονείς τους για τα ψηφιακά ή και περισσότερα. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα είδη πόρων για καθοδήγηση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλες οι πηγές. Ήταν πολύ θετική η εμπειρία μας. Χρησιμοποίησαμε ένα σύστημα ταξινόμησης περιεχομένου. Υπάρχουν πάρα πολλές γνώσεις για το θέμα αυτό. Και θεωρείται αυτό ένα εργαλείο καθοδήγησης εξαιρετικά αποτελεσματικό η επένδυση στην καθοδήγηση των γονέων είναι καθοριστικό, είναι βασικό. Και αυτό πρέπει να επεκταθεί να, για να αφορά όλο το περιεχόμενο, γιατί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το περιεχόμενο είναι απολύτως επίκαιροι. Ευχαριστώ. Για να προσθέσω σε σχέση αυτό που έλεγε ο Μπράιαν, Πράγματι χρειαζόμαστε γονείς με περισσότερη εμπειρία, ε, με περισσότερες γνώσεις. Η αλήθεια είναι ότι όσοι γονείς είναι από τα υψηλότερα, να το πω έτσι, κοινωνικά στρώματα, είχαν περισσότερες γνώσεις. Οι γονείς από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα περιορίζουν την πρόσβαση. είδαμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι με την υπερχρήση και την ανεξέλεγκτη χρήση της ψηφιακή τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει στα δικοκυριά όπου οι γονείς δεν έχουν χρόνο. Δεν είναι θέμα πόρων στην οικογένεια, αλλά έλλειψη χρόνου. Οι γονείς δεν ε, περνούν αρκετό χρόνο με τα παιδιά τους δεν είχαν χρόνο να δουν πώς τα παιδιά τους χειρίζονται στη τεχνολογία και μάλιστα μερικές φορές την ενθαρρύνουν και αυτή τη χρήση γιατί η ψηφιακή τεχνολογία είναι πιο ασφαλής ή έτσι να αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι είναι πιο ασφαλής από πλευρά σώματος για τα παιδιά, δηλαδή δεν κινδυνεύει το σώμα αυτό καθεαυτό. Είναι σαν να έχει το παιδί μια ψηφιακή babysitter και δεν κινδυνεύει να χαθεί ή οτιδήποτε τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άρα τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη των ε, ε, σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που καλούνται ακριβώς να αντισταθμίσουν ή να εξισορροπήσουν τα όσα δεν προσφέρονται ή δεν μπορούν και να προσφερθούν στο σπίτι. Περνάμε λοιπόν στο στο δεύτερο, στο δεύτερο γύρο. Ε, η κυρία Στίβενς έχει το λόγο. Uh, Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την μελέτη που εκπώνησα. Εξετάσαμε διάφορα νομοθετικά ρυθμιστικά εργαλεία για την ε, πλαισίωση των δικαιωμάτων του παιδιού στην ψηφιακή εποχή λύσεις αλλά και διλήμματα πολιτικής. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι τον σεβασμό των ε, δικαιωμάτων του παιδιού ε, υπάρχουν ήδη μια σειρά από ε, εργαλεία. Η νομοθεσία, η αποκοινού ρυθμίση και η αυτορύθμιση έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να δημορφωθεί το, το πλαίσιο, το περιβάλλον. Και εδώ υπάρχουν διάφορα επίπεδα συμμετοχής ε, των επιμέρους φορέων και παραγόντων. Για παράδειγμα, στην, στην νομοθεσία, στο δίκαιο, προφανώς ε, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, ε, στην, ε, στην, στην αυτορύθμιση παίζουν ρόλο κυρίως οι επιχειρήσεις και η αποκοινού ρύθμιση βεβαίως περιλαμβάνει τις δύο αυτές πλευρές, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν είναι πολύ σημαντικά, ακριβώς γιατί αποτελούν και ένα συνεχές, μια συνέχεια. Και παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυτορύθμιση, υπάρχει μια μετάβαση ε, σε μια ε, πιο προηγμένη μορφή από κοινού ρύθμισης πλέον. Οι πρόσφατες ε, νομοθετικές πράξεις, όπως είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ή ε, η οδηγία για τα οπτικοστικά μέσα ε, δείχνουν ακριβώς αυτό. Και παρά το γεγονός ότι τα νομοθετήματα αυτά ε, προβλέπουν πιο αυστηρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Και αυτό, αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, γιατί ακριβώς αφενός συνδυάζει αυτή η από ρυθμίση και την ε, εποπτεία, τη δημοκρατική λογοδοσία, αλλά και την ε, ε, προαγωγή των τεχνολογικών εξελίξεων. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα, απαραίτητα στοιχεία είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός. Ταυτόχρονα πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων σε όλα τα δικαιώματα του παιδιού. Υπάρχει για παράδειγμα και το, το, το, το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης ή της ιδιωτικότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναγνωριστεί ότι διάφορες, διαφορετικές ηλικίε χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία. Και βεβαίως να μην ε, υπερτιμούμε και την αποτελεσματικότητα της ε, τεχνολογίας. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία επαλήθευσης ηλικία ε, προκειμένου να επιβάλλονται περιορισμοί σε συγκεκριμένα είδη περιεχομένου στα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση τα παιδιά, όπως είναι σεξουαλικό περιεχόμενο ή ε, ιστοσελίδες τζόγου. Υπάρχουν διάφορες μεθόδους, ε, μέθοδοι που μπορείς να χρησιμοποιήσει κανεί, όπως είναι έλεγχοι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να υπερρυθμίζεται, να ρυθμίζεται υπερβολικά ε, αυτό το θέμα. Γιατί ε, η, η, η ελάχιστη χρήση δεδομένων, η ελάχιστη δυνατή χρήση δεδομένων, όπως ορίζει και ο κανονισμός, είναι αυτό που πρέπει να είναι το, το ζητούμενό μας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες στρατηγικές για την αύξηση και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά δεν είναι και πανάκια. Αυτό χρειάζεται ταυτόχρονα εκτός από την ε, την αύξηση των δεξιοτήτων, να υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και η αυτορύθμιση από τις επιχειρήσεις. Το να δίνεται λοιπόν η δυνατότητα αυτή στους γονείς, ε, όπως ε, τα συστήματα αξιολόγησης, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ένα βασικό στοιχείο στην νομοθετική διαδικασία. Αν λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο η στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού στο στην ψηφιακή εποχή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, τότε βεβαίως ανακύπτουν διάφορα διλήμματα. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα τα δικαιώματα των, των παιδιών, προστασία, συμμετοχή και πρόληψη, πρέπει να καθοδηγούν την νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα ζητήματα πολλές φορές επικαλύπτονται, κάποιες φορές μάλιστα συγκρούονται κιόλα. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα του παιδιού ε, στην ε, ε, ελευθερία παραλαβής ε, πληροφοριών και ενημέρωσης μπορεί κάποια στιγμή να συγκρούεται με το δικαίωμα τους να προστατεύονται από επιβλαβές περιεχόμενο όπως το περιέγραψε ο Μπράιαν. Άλλες περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις, περιορισμός στη χρήση τεχνολογικών μέσων σε σχολεία, δήμους ή βιβλιοθήκες δεν είναι τόσο ε, σημαντική και έτσι εκεί μπορεί να γίνει προσβάσιμο αυτό το ακατάλληλο περιεχόμενο. Περιορισμοί λοιπόν χρειάζονται, πρέπει πάντοτε να είναι, να είναι αναλογικοί όμως, ουσιαστικοί και να εξυπηρετούν τον ε, βασικό μας στόχο, την προστασία. Επίσης, ε, σημαντικό είναι και ε, η εκάστοτε ηλικιακή ομάδα για την οποία καταρτίζουμε έναν περιορισμό ή έναν κανόνα. Συγκρούσεις λοιπόν μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ μεγαλύτερων παιδιών, εφήβων, τα σεξουαλικά του δικαιώματα και την προστασία, το δικαίωμα της προστασίας τους. Ή ζητήματα όπως είναι το sexting. Η ποινικοποίηση λοιπόν κοινή χρήση ε, σεξουαλικών εικόνων ε, σε ε, εθελοντική βάση μεταξύ εφήβων και ο περιορισμός αυτής της δυνατότητας μπορεί να αποτελεί και παραβίαση του δικαιώματός τους στην συγκρότηση της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Άρα πρέπει οι φορείς χάραξης πολιτικής να ε, φύγουν από μια προσέγγιση ε, κατασταλτική, περιοριστική και να ενθαρρύνουν την, ε, την αυτορύθμιση. Γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η ενίσχυση του δικαιώματος να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό τους και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και επίγνωση των προβλημάτων των κινδύνων που ενέχονται στο διαδίκτυο. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ε, ο στόχος προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων των παιδιών δεν πρέπει να υπονομεύει το δικαίωμά τους στη συμμετοχή. Έχει ε, Υπάρχει, λοιπόν ο ισχυρισμό ότι το άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες, διάφορες υπηρεσίες να μην προσφέρουν τα, προϊόντα τους σε ε, μικρά παιδιά ακριβώς γιατί δεν θέλουν να περιπλέξουν την, ε, τις δικές τους διαδικασίες και το να πρέπει να πάρουν συγκατάθεση διαρκώς από τους γονείς. Αυτό όμως μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα στο παιχνίδι των παιδιών. Επιπλέον, κατά τη χάραξη ρυθμιστικών πολιτικών, η πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οι ευθύνε μια σειρά φορέων και εμπλεκομένων όλοι οι παράγοντες εδώ που βλέπετε, σε αυτή τη διαφάνεια, φέρουν σε κάποιο βαθμό κάποιες ευθύνες. Αν και ε, το, το, το ποιες ευθύνες και σε ποιο βαθμό αναλογούν στον καθένα είναι ζήτημα που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί οριστικά. Πάντως, σε έναν ε, συνδεδεμένο κόσμο, η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της βιομηχανίας ε, και των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι θετικό. Πρέπει λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία να, να εμπλέκονται και να συμμετέχουν και οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών, όλοι οι εμπλεκόμενοι και να υπάρχουν σαφείς στόχοι, σαφείς, σαφείς συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης, ασφαλιστικές δικλείδες. Και όταν υπάρχει επικοδομητική συνεργασία μεταξύ ρυθμιστών και ρυθμιζομένων, τότε ε, επιτυχάνονται τα καλύτερα ε, αποτελέσματα. Οι φορείς που ε, πρέπει να εμπλακούν περισσότερο ε, στο μέλλον είναι τα παιδιά και η κοινωνία των πολιτών. Τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν στη χάραξη και τη διαμόρφωση πολιτικών που θα διαμορφώσουν και το ψηφιακό περιβάλλον εντό του οποίου ζουν ε, και χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη δική τους φωνή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θετική ε, τάση. Ε, υπάρχει η αποκοινή, αποκοινού ρύθμιση δηλαδή η συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, με ευελιξία αλλά και με παρακολούθηση, και το βλέπουμε αυτό στι εξελίξει, για παράδειγμα, όσον αφορά τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων και την Οδηγία για τι Οπτικοακουστικές υπηρεσίε. Επίση, υπάρχει μια τέτοια θετική τάση, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιώματα του παιδιού και να μην δίνεται υπερβολική έμφαση μόνο στην πλευρά τη προστασία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, υπό το φως των συστάσεων που θα εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης πολύ πρόσφατα. Και εκεί λοιπόν υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα δικαιώματα του παιδιού. γιατί ακριβώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιώματα των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και την ηλικία τους, αλλά και τις καταστάσεις εντός των οποίων ενδέχεται να βρεθούν τα παιδιά. Και Τέλος, συμφωνώ με τη σύσταση του Μπράιαν ότι όλες οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε ενδείξεις, σε στοιχεία που θα παρακολουθούν τις εμπειρίες των παιδιών όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό βεβαίως χρειάζεται πόρους και εντολή προκειμένου να διεξάγονται οι αντίστοιχες έρευνες και μελέτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι φορείς χάραξης πολιτικής επίσης θα πρέπει να εξετάσουν ε, και το ενδεχόμενο να, να, να διεξάγονται επί τούτου μελέτες αντικτύπου για τα δικαιώματα των παιδιών πριν από τη χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής και την υποβολή οποιασδήποτε νομοθετικής πρότασης. Αυτό Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέτοιου είδου αξιολογήσει αντικτύπου πρέπει να διεξάγονται πάντοτε και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε για τι εκτιμήσει σα. Μα καθιστούν σαφές το δίλημα, τα διλήμματα ενώπιον των οποίων βρίσκονται και οι πολιτικοί. Θα επανέλθουμε βεβαίω, αλλά πρώτα περνάμε στην τελευταία μα παρουσίαση τη κυρία Λίβινγκστον. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας απευθύνω τις προτάσεις και συστάσεις μας σήμερα. Συνεχίζω στα όσα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι για τη διατύπωση των συστάσεων. Είμαι καθηγητρία στο London School of Economics. Εξετάζω κυρίως τα θέματα των ε, παιδιών και των ευκαιριών, ιδιαίτερα σε σχέση με το διαδίκτυο και τα δικαιώματα των παιδιών ε, και έχω ασχοληθεί με τα θέματα χάραξης πολιτικής. Μια έκθεση λοιπόν που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα, την έχουμε επεξεργαστεί με δύο συναδέλφους ειδικού στα θέματα των ε, μέσων μας και ενημέρωσης και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα σας εξηγήσω τα τρία καθήκοντα τα οποία εντοπίζω για την έκθεση αυτή, δηλαδή τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αξιολόγηση των υφισταμένων πρωτοβουλίων και εργαλείων και τη διατύπωση συστάσεων προς την Επιτροπή σας για περαιτέρω εξελίξεις. Επομένως, σε τι πλαίσιο κινούμαστε, βρισκόμαστε, όπως υπόθηκε ήδη νωρίτερα σήμερα, σε ένα περίπλοκο σύστημα προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, με νομοθετικές ε, ε, παρεμβάσεις και αυτορύθμιση, ε, που ωστόσο δεν προχωρεί τόσο γρήγορα όσο το περιβάλλον το ψηφιακό και αντίστοιχα οι κίνδυνοι για τα παιδιά. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός χάρτη ε, του χάρτη για τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του χάρτη για τα δικαιώματα των παιδιών. Ιδιαίτερα απαιτούνται κοινέ προδιαγραφές, κοινά πρότυπα και όπως ε, κατέστησε σαφές και ο Μπρέν ο Νίλ νωρίτερα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, με πολλές ενδείξεις για βλάβη εις βάρος των παιδιών, παρά τις πολλές προσπάθειες για προστασία τους και αυτό γιατί είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ε, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Είναι πολλοί, πολλαπλοί οι κίνδυνοι που ελοχεύουν ε, στο διαδίκτυο για τα παιδιά και είναι όλο και πιο δύσκολο να προληφθούν, να προβλεφθούν είναι πολύ δύσκολο και ε, να αντιμετωπιστούν ή να δοθούν λύσεις γιατί είναι πολλοί οι διάφοροι φορείς που εμπλέκονται στην εξασφάλιση λύσεων. Από το 12 λοιπόν που είχαμε κάνει μια διεξοδική χαρτογράφηση των προβλημάτων και με φραγμούς που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνη για τη χάραξη πολιτικής. Κάποιες ε, ολίγες καλές συστάσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Εγώ θα προσπαθήσω να αξιολογήσω τις πρόσφατες εξελίξεις και να διατυπώσω νέες συστάσεις. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική από το 2012, από την τελευταία μας έκθεση. έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτορύθμιση, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενημέρωση Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολέμηση της σεξουαλικής δαπαρινόξης ε, διαδικτυακά για τα παιδιά έχει επίσης πάρει μεγάλη έμφαση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε περισσότερο την ενιαία ψηφιακή αγορά και τη στην ε, πρόσφατη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αυτής στρατηγική, Τα παιδιά δεν αναφέρονταν σχεδόν καθόλου, παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον και επίση δεν υπάρχουν αρκετέ συστάσει, συγκεκριμένε συστάσει για την προστασία των παιδιών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξελίξη λοιπόν από το 2012 σε σχέση με την νομοθεσία έχουμε ένα κανονισμό γενικό, προστασία προσωπικών δεδομένων, καλύφθηκε ήδη από την προηγούμενη ομιλήτρια. Ε, στην αυτορύθμιση έχουμε μια συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων ε, διαγραμμικά, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο δίκτυο προστασίας για τα παιδιά ή καλύτερο διαδίκτυο μάλλον για τα παιδιά και αναθεώρηση της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές ε, υπηρεσίες η οποία προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και βέβαια εισάγει λύσεις για αυτά που το Κοινοβούλιο καταγγέλει ως ρυθμιστικές αποτυχίες. Κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία της έκφρασης. Ε, Θέλετε να μιλάτε λίγο πιο γρήγορα για να σας παρακολουθούμε πιο καλά. Α, ναι, με συγχωρείτε. Άλλες λοιπόν ε, κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία της έκφρασης διαδικτυακή ε, επιμόρφωση, επιμόρφωση στη χρήση των μέσων, καταπολέμηση του, της ρητορικής του μίσους που μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την συνρύθμιση. Ναι, ειδικά όταν διαβάζουν οι ομιλητές χωρίς να δώσουν. Μπορείτε να δώσετε το έγγραφο στους ε, διερμηνείς αν έχετε την καλοσύνη. Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο από τον αρχίσετε από την αρχή. Το καθεστώς λοιπόν για την ευθύνη του ενδιάμεσου θεμελιώδη δικαιώματα για τα παιδιά που δεν έχει αλλάξει από το 2012, συνεχιζόμενες συζητήσεις, ανησυχίες που εξακολουθούν να εκφράζονται, αδυναμία και αδικία του να περιορίσετε το παιδί σε έναν ε, κήπο με ψηλού στίχου σημαίνει ότι η πρόκληση είναι μεγάλη και για το, την προστασία του παιδιού αλλά και για τον ρυθμιστή που θέλει να εξασφαλίσει ένα ψηφιακό περιβάλλον για όλους. Επομένως ένα καλύτερο ε, πλαίσιο και πάνω απ' όλα καλύτερα συντονισμένο πλαίσιο και νομοθετικό αλλά και κινήτρων μπορεί να είναι η σωστή λύση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις καταγράφει, υπάρχουν και διεθνείς προσπάθειες ε, όπως από την Ένωση, Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών, ε, Παγκόσμια Συμμαχία, Συμμαχία ε, Κοινωνίας Πληροφορίας για τα Δικαιώματα των Παιδιών κ.ο.κ. στην αξιολόγηση των υφισταμένων πρωτοβουλειών και μέσων ή εργαλείων. Μεγάλο κομμάτι της εκθεσής μου σας έχω βάλει φωτογραφίες παιδιών που χρησιμοποιούν την ε, ψηφιακή τεχνολογία στο σπίτι, στο σχολείο ή αλλού. Και αυτό μας θυμίζει ποιος είναι τελικά ο αποδέκτης των προσπαθειών αυτών, ποιος πρέπει να ωφεληθεί από τις προσπάθειες αυτές. Άρα πρέπει και τις απόψεις των παιδιών, των δασκάλων αλλά και των γονέων να συλλάβουμε υπόψη για να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πολλά είναι λοιπόν τα προβλήματα, οι δυσκολίες σχέση με τα εργαλεία αξιολόγησης, ε, έννοιες που πολλές φορές ε, δεν είναι κατανοητές, η εργαλεία που δεν είναι γνωστά στους γονείς και τα παιδιά, ε, ευθύνες που δεν μπορεί να γνωρίζουν ακριβώς, η δυσφορία που αισθάνονται, η ανησυχία γιατί βλέπουν ότι δεν ανταποκρίνεται το ψηφιακό περιβάλλον στις προσπάθειές τους. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν απαντά ούτε στις ανάγκες τους ούτε στις ε, ανησυχίες τους και δεν δίνει απαραίτητα και τα εργαλεία που χρειάζονται. Τόσο γονείς σου και παιδιά συχνά αισθάνονται σύγχυση ως προς τις ε, ε, διαφορετικές προσεγγίσεις διαφορών ε, επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικά εργαλεία, επιλογές, προτιμήσεις και έτσι συχνά λένε ότι δεν εξασφαλίζουν ε, στις έρευνές μας, δεν εξασφαλίζουν τα εργαλεία που θέλουν και ότι, δεν υπάρχει, και ότι υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να ξεφύγουν από τα εφιστάμενα συστήματα προστασίας. Βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο ε, δραστηριότητες με πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς ε, μπορούν να δώσουν ε, κάποιες απαντήσεις ως προς τη διευκρίνηση των καθηκόντων και των ευθυνών των παρόχων υπηρεσιών σε όλη τη διαδικασία και την αλυσίδα. Σημαντικό επίσης είναι να μην είναι ανεπαρκής η παρακολούθηση και η επαλήθευση της συμμόρφωσης, δηλαδή τα στοιχεία της αποτελεσματικότητας. Είναι πολύ δύσκολο να τα αναγνώσουμε. Ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα παιδιά είναι αυτά που θα χαθούν κάπου στη διαρεύνηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας να κάνουμε τις ερευνές μας. Και έτσι καταλήγω σε κάποιες συστάσεις. Συνιστούμε η στρατηγική για το καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά να αναπτύξει έναν πλήρη κώδικα βέλτιστης συμπεριφοράς, άριστης συμπεριφοράς, ε, με οδηγίες για τους παρόχους υπηρεσιών ε, διαγραμμικών για τα παιδιά που θα πρέπει να ενσωματωθεί ή δυνατόν στο σχεδιασμό των υπηρεσιών και εργαλείων, δηλαδή ιδιωτικότητα, ιδιωτικός βίος, σχεδιασμός, ε, στόχευση με τα συμφέροντα του παιδιού σαν κύριο γνώμονα, σαν πρωταρχικό και κύριο γνώμονα. Όλο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα της ανάσχεσης, ισχυρές εξουσίες ανάσχεσης, ανεξάρτητης παρακολούθησης και αξιολόγησης. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δίνει καθοδήγηση για τους ενδιαμέσους τις διαδικασίες και τις ευθύνες που έχουν για την προστασία του παιδιού, να δίνει σαφείς πληροφορίες για την προστασία του καταναλωτή και σημεία προστασία εάν οι υπηρεσίες δεν στοχεύουν τα παιδιά. Δεν επιτρέπεται να ε, γίνει χρήση του από τα παιδιά. Και βέβαια αντίστοιχα θα πρέπει να προωθηθούν και οι καλύτερες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών. Για να είναι αποτελεσματικός αυτός ο κώδικας θα πρέπει να έχει και επαλήθευση ηλικία και άλλα φίλτρα και δυνατότητα κλεισίματος ή κατεβάσματος. Θα μπορούσε να έχει έναν κατάλογο συνιστομένων υπηρεσιών ή διαδικτυακών ε, πόρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί άφοβα ε, το σχολείο, για το σχολείο του, για τους γονείς του, ε, ελάχιστες προδιαγραφές που επίσης αντίστοιχα αν δεν γίνονται σεβαστές θα οδηγούσαν σε απάλληψη από τον κατάλογο, το θετικό αυτό κατάλογο. Συστάσεις επίσης, συνεχίζω, μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προήγαγε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ψηφιακή γνώση, ε, με τη δυνατότητα παραγωγής πρόσθετων δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, που θα επικαιροποιείται διαρκώς όσο εξελίσσεται, όπως εξελίσσεται και το σχετικό περιβάλλον και θα επιτρέπει την προσαρμογή και όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας του εκπαιδευτικού συστήματος, ε, γενικότερα της συμμετοχής σε θελοντική βάση και βέβαια η οδηγία για τα οπτικοακουστικά θα έχει κρίσιμη και ζωτική σημασία και θα πρέπει να προβλέψει και μια δραστηριότητα παρακολούθησης της εφαρμογής. Συντονισμό επίσης συνιστούμε σε επίπεδο ομάδας αξιωματούχων υψηλού επίπεδο και σε, μόνιμο, σε μόνιμη επιτροπή με την παρακολούθηση του κώδικα, της σύστασης, και της αξιολόγησης ε, μέτρων ε, των κρατών μελών που μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμα ε, και έτσι να συνδυάζονται και οι δράσεις και να εξασφαλίζονται κοινέ προδιαγραφές και πρότυπα μέσα σε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να αξιολογείται ανεξάρτητα, να έχει υποχρέωση λογοδοσίας, να είναι ουδέτερο. και εν τέλει Οι συνάδελφοι ανέφεραν, ανέφεραν τη σημασία της χαράξης πολιτικής με βάση στοιχεία και δεδομένα στέρεα. Βεβαίως θα πρέπει τα παιδιά να είναι σε θέση να εκφραστούν σε θέματα που όπως το συγκεκριμένο τα αφορούν άμεσα για να ολοκληρώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πάρα πολλά για να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Υπάρχουν όμως ακόμα σοβαροί κίνδυνοι και σοβαρή βλάβη στα βάρο των παιδιών. Υπάρχει ο κίνδυνος της κλιμάκωση της επικινδυνότητας και ύστερα από τόσα χρόνια που έχουν, που έχουν αναλυφθεί δράσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, ακόμα πολλά μένουν να γίνουν. Επομένω, το Κοινοβούλιο πρέπει να ε, θεσπίσει και να εισαγάγει σαφεί προδιαγραφέ, να επιτρέψει την συμμετοχή σε διαδικασία δικασίες πολλών ή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να είναι σαφές και για την αγορά τι μπορεί να περιμένει, αλλά και να είναι σαφείς οι προδιαγραφές και οι κώδικες. Και επίσης υπόθηκε νωρίτερα ε, και λέγεται συχνά, σπάνιο όμως εφαρμόζεται στην πράξη, δράσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό, για την ε, εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να είμαστε θέσει να προλάβουμε τα περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και περνάμε τώρα στην επόμενη, ε, στον επόμενο γύρο συζήτηση. Σίλβια Κώστα. Προσπάθησε παρακαλώ σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και βεβαίω θέλω να πω ότι τα σημερίζομαι. Το ψηφιακό περιβάλλον σήμερα είναι το νέο όριο των δικαιωμάτων των παιδιών και των ε, εφήβων. Ωστόσο, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει μια εγκάρσια προσέγγιση ομοιόμορφη ακόμα και στην ψηφιακή στρατηγική. Υπάρχουν επιμέρους λύσεις, αλλά όχι συνολικά. Επιμέρους λύσεις είναι και για την ιδιωτικότητα, για την προστασία του ιδιωτικού βίου και για τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει μια ολιστική, μια εγκάρσια προσέγγιση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο πράγματα θέλω να πω, ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου μπορεί η νομοθεσία και ε, ατελής έστω να δίνει ε, λύσεις αλλά και να συνυπάρχει με κώδικες αυτορύθμισης, δηλαδή ρύθμιση και συρρύθμιση, ε, διαδικασίες ε, η παρέμβαση των αρχών και όμως εδώ πρέπει να δούμε την δίωξη της κυρώσης που είναι απαραίτητες, αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα και βεβαίως υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι δεν έχουν καλυφθεί και είναι τέρα ε, incognita. Εγώ θα ήθελα να δω λοιπόν εάν ε, τα κράτη, που όπως άλλωστε προτείνει και η οδηγία μας δίνει την επιλογή περισσότερο στον ιδιώτη. Αυτό όμως προβλέπεται ήδη σε εμπορικό επίπεδο, άρα πρέπει να δούμε κάποιες διαφορετικές λύσεις. Και οι αρχές οι αρμόδιες, οι παραδείγματι στη χώρα μου, έχουμε μία ένα σώμα αστυνομικό, μια μονάδα της αστυνομίας που ασχολείται μόνο με το κυβερνοέγκλημα και πιστεύω ότι, θα είναι, ότι είναι μια καλή ιδέα και θα έπρεπε να διαδοθεί και σε άλλες χώρες. Επίσης, ο κυβερνοεκφοβισμός cyberbullying και στη χώρα μου έχει εισαχθεί ένα ενδιαφέρον νομοθέτημα πρόσφατα. Να, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια ιδέα ή σχόλιο, αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και επίσης, για να ολοκληρώσω... Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά εγώ πάντως πιστεύω και καταγράφω ότι πρέπει, θα έπρεπε να υπάρχει ένας κώδικας ε, καλής συμπεριφοράς πιο εκτεταμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινό ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως θα μπορούσαμε και να εξασφαλίσουμε από την έργα την καθοδήγηση με την καταγραφή των ελάχιστων προδιαγραφών και ταυτόχρονα... Ναι, ναι, ναι τελειώνω. Ε, περισσότερη έμφαση στο ρόλο του ενδιαμέσου, του διαμεσολαβητή στην χρήση του ψηφιακού περιεχομένου. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κύριε Μπίλτ. με συγχωρείτε. Έχουμε πινκ-πονγκ τώρα, ναι. Επομένως, πρώτα θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις αυτές. Ένα από τα βασικά ζητήματα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο είναι ότι είναι πολύ διαφορετικές οι αρμοδιότητες, οι αρμόδιοι φορείς. Άλλο Υπουργείο είναι αρμόδιο για κάποιο θέμα σε ένα μέρος, άλλο Υπουργείο είναι αρμόδιο σε άλλο. το γεγονός ότι η ζωή των παιδιών κυριαρχείται από την τεχνολογία και είναι ουσιαστικά βεθισμένα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον σημαίνει ότι υπησέρχονται θέματα υγείας, θέματα μέσων μαζικής επικοινωνίας, θέματα τεχνολογίας, πολλά και διάφορα. Δεν είναι αρκετός ο συντονισμός. Για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα Υπουργεία καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες και ότι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Περισσότερο συντονισμός. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Και η ιδέα του κώδικα δεοντολογίας θα καταλάγιαζε τις αβεβαιότητες. Πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς νιώθουν εξαιρετικά αβέβαιοι. Ε, και το ανέφερε και η Σόνια. Και τα παιδιά και οι γονείς δεν ξέρουν τι να περιμένουν από ορισμένε υπηρεσίες. Δεν ξέρουν αν το YouTube υπάγεται στους κανόνες της τηλεόρασης, αν υπάγεται σε οποιουσδήποτε κανόνες. Αλλά και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται γιατί πρέπει να εκπληρώσουν και να σταθούν στο ύψος πολλών και διαφορετικών υποχρεώσεων. Επομένως, ένα εργαλείο συντονισμού, ελάχιστα πρότυπα και κώδικας διοντολογίας δηλαδή, ε, θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό και χρήσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η Σόνια Λίβινγκστον παρακαλώ. Συμφωνώ και εγώ με τη σειρά μου. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε ένα μείγμα εργαλείων και πρέπει να καταλήξουμε στο σωστό μείγμα. Αλλά θα πρέπει να τυποποιήσουμε και να δώσουμε ε, σάρκα και οστά σε αυτό το χαοτικό πεδίο, να το κατατάξουμε κάπως και να το οργανώσουμε. Πρώτον, μιλούμε για τις ε, ευθύνες των ενδιάμεσων της κάθε πλατφόρμας και εκεί πρέπει να έχουμε ελάχιστα πρότυπα που ε, καθορίζονται και από τον κώδικα δεοντολογίας. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί τα παιδιά και οι γονείς, άρα πρέπει να ε, κάνουμε σημαντικές προσπάθειες για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τρίτον, συντονισμό των ευθυνών μεταξύ γονιών και παιδιών και των ευθυνών των κυβερνήσεων και των εταιριών σε σχέση με το κώδικα δεοντολογίας. Χρειάζεται μια ομάδα συντονισμού για όλα αυτά που θα δραματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά και οι συστάσεις είναι πολύ σημαντικές. Δεν θα φύγει αυτή η πρόκληση. Ε, δεν πρέπει να είναι προσωρινή αυτή η ομάδα να έρθει να φτιάξει τα πράγματα για κάθε χρόνο και να φύγει. Πρέπει να είναι μια μόνιμη ομάδα συντονισμού, γιατί όσο εξελίσσεται η τεχνολογία θα προκύπτουν και νέες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη ομάδα εποπτείας παρακολούθησης που να έχει μάλιστα σημαντικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ευχαριστώ κυρία Μπίλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω κι εγώ να μιλήσω αργά. Είναι επίγον να βρούμε νόμιμες λύσεις στις καταχρήσεις του διαδικτύου. Υπάρχουν ήδη αυτές οι λύσεις στο ποινικό δίκαιο. Να σημειώσουμε ότι το πιο πιεστικό πρόβλημα για τα θύματα είναι να καταφέρουν να διατηρήσουν και να διασώσουν και να προφυλάξουν την εικόνα και την προσωπική του ζωή στο διαδίκτυο. Για να αποφύγουμε αντίκτυπο μακροπρόθεσμο στην επαγγελματική και προσωπική ζωή σε σχέση με το πόσο κρατούν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο το 80% των εργοδοτών που προσλαμβάνουν χρησιμοποιούν το Google για να μάθουν πράγματα για τον άνθρωπο που θέλουν να προσλάβουν. Και μπορεί αυτό να στοιχήσει μια φωτογραφία πριν από πολλά χρόνια να στοιχήσει τη δουλειά ή να μην μπορέσει κάποιος να νοικιάσει σπίτι γιατί ο ιδιοκτήτης το έχει ψάξει και είδε πράγματα που δεν του αρέσουν ε, πάρα πολλά χρόνια πριν δεν έχουμε το δικαίωμα στη λύθη. Υπάρχει το, ο κανονισμός του 2016 και έτσι αυτό θα ρυθμίσει. Είναι νομική βάση για τους ανηλίκους που ήταν θύματα εκφοβισμού, παρενόχλησης που έχουν διαδοθεί εικόνες χωρίς την άδειά τους έτσι ώστε να προστατευτούν καλύτερα. Έχουμε ε, ε, επιδόσεις φρικτές σε ορισμένες χώρες και υπάρχουν Και υπάρχει και η περίπτωση της Τιτσιάνα Καντόνε ε, που τελικά ε, οδηγήθηκε στο να χάσει ε, τη ζωή της. Έχουμε περιστατικά δηλαδή σε χώρες πραγματικά φρικτά ακριβώς γιατί δεν υπήρχε αυτό το δικαίωμα στη λύθη. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Αν δούμε το κανονισμό, το άρθρο 17 γιατί γενικότερα η προστασία των δεδομένων, πράγματι το δικαίωμα στη λύθη, στη διαγραφή, έχει αναφερθεί πολύ ρητός, έχει αναφερθεί ως εξαιρετικά χρήσιμο στα παιδιά που έχουν αποκαλύψει δεδομένα και στοιχεία στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά έχετε δίκιο. Πρέπει να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Καταρχάς, για να το ασκήσουν αυτό το δικαίωμα τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι το, πρέπει να μάθουν ότι το έχουν. Άρα περισσότερη εκπαίδευση για τα δικαιώματα, για την προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί κανείς να ασκήσει ένα δικαίωμα τα οποία δεν γνωρίζει ότι έχει. Επίσης, στην πράξη, η αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Άρα χρειάζονται καθοδηγήσεις, κατευθυντήριες γραμμές από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων για να ενημερώσουν τους ελεγκτές για θέματα περιεχομένου πώς θα το πράξουν αυτό. και να είναι εξαιρετικά πιο προσεκτικοί, πολύ πιο προσεκτικοί όταν ξέρουν τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν παιδιά. Βεβαίως, συμφωνώ και με αυτό που είπατε στην αρχή. Χρειάζεται ποινική νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις. Να εφαρμοστεί αυτή. Για παράδειγμα, διάδοση εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς την συγκατάθεση. Όλο και περισσότερες χώρες το ποινικοποιούν αυτό. Τα παιδιά πρέπει να το γνωρίζουν ότι δεν είναι ποινικό επιτροπτό να ε, διαδίδει κανείς χωρίς ή κατάθεση εικόνες ε, με σεξουαλικό περιεχόμενο και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην εκπαίδευση για τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και την εκπαίδευση ε, για τη σεξουαλική αγωγή και για τη σημασία της συγκατάθεσης γενικότερα. Η κυρία Λίβιγκστον, είναι πολύ σωστά τα ερωτήματά σας και θα ήθελα να προσθέσω κάτι στα λεγόμενα της ΕΒΑ Δύσκολο να φανταστούμε μια Ευρώπη όπου τα παιδιά θα ασκούν αγωγή στις επιχειρήσεις για να πάρουν πίσω τις εικόνες τους και το περιεχόμενό τους από τις επιχειρήσεις φυθιακού περιεχομένου. Θα πρέπει να είναι αυτό το τελευταίο μας καταφύγιο, να έχουμε κανόνες και εξέλιξη στην νομοθεσία και στις ε, ε, στα μέτρα που να μας ε, κάνουν να αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κώδικας διοντολογίας σε θελούσια βάση θα αλλάξει ε, με κάποιο τρόπο το σχεδιασμό των υπηρεσιών έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι και να μην καταλήξουμε σε πόλεμο μεταξύ παιδιών και επιχειρήσεων. Γιατί ο πύχης της δικαιοσύνης είναι πολύ υψηλός για να μπορέσουν να το φτάσουν τα παιδιά Το σημαντικό είναι να θέσουμε συγκεκριμένα πρότυπα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ε, προτύπων ε, συμπεριφοράς από πλευράς χρηστών. Μιλούμε και για χρήστες παιδιά, αλλά και για ενήλικες, χρήστες ενήλικες. Τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα χώρο ε, στον οποίο μπαίνουν μόνο παιδιά. υπάρχουν πολλοί ενήλικοι που συμπεριφέρονται με προβληματικό τρόπο στη διαδικτυακή τους ζωή. Άρα πρέπει να αλλάξουν και κάποια πρότυπα συμπεριφορών που γίνονται ανεκτά. Δεν λέω ότι θέλουμε μια προσέγγιση λογοκρισίας, αλλά πρέπει να βρούμε κάποια λύση για να έχουμε μια συμπεριφορά πιο πολιτισμένη με περισσότερο σεβασμό στον συνάνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, Julie Ward. Σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Δεν ήμουν από την αρχή, όμως νομίζω ότι αποδεικνύει το σημερινό εργαστήριο τη σημασία που, έχουν, που έχει διοργάνωση τέτοιου είδους εργαστηρίων από τους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι ακούσαμε από σας την οπτική των δικαιωμάτων των παιδιών. Νομίζω ότι η θέση των παιδιών έχει υποβαθμιστεί στις κοινωνίες μας. Η λιτότητα σημαίνει περικοπές δαπανών για τα παιδιά, για κέντρα και συλλόγους που ασχολούνται με την απασχόληση των παιδιών. Η αδερφή μου είναι ε, δασκάλα και μου έχει πει ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι στο σχολείο της είναι σαν να τις λένε από το Υπουργείο κάντε αυτά, αλλά όχι ότι δίνουμε και ιδιαίτερη αξία στην, ε, στο επάγγελμά σας ή στην, στη ζωή του παιδιού. Γονείς αναγκάζονται να κάνουν μία, δύο, τρεις, τέσσερις δουλειές κάποιες φορές. Άρα πρέπει να δούμε πώς η λιτότητα έχει επηρεάσει αρνητικά αξίες που μοιραζόμαστε όλοι, όπως είναι η προστασία των παιδιών. Και επειδή είμαι Βρετανίδα και με ανησυχεί πάρα πολύ το Brexit και ε, συνεργάζομαι με οργανώσεις προστασίας των παιδιών που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σε ένα όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποια είναι η αίσθηση και τι προβλέπετε εσείς ε, εν ώψη του Brexit ε, και δεν εννοώ μόνο για το τι θα συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, ε, ποιε θα είναι και οι επιπτώσει στι άλλε 27 χώρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λίβινγκστον. Ανησυχώ και εγώ πολύ. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μόνος φορέας αυτή τη στιγμή που έχει την εμπειρογνωμοσύνη, την εξουσία αλλά και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει τη δύναμη των μεγάλων εταιριών που με πολλούς τρόπους σχεδιάζουν τα προϊόντα στα οποία εμείς ε, βγάζουμε τη ζωή μας ε, ή γύρω από, τις οποίες, γύρω από τα οποία οργανώνουμε τη ζωή μας, όπως είναι τα social media για παράδειγμα. Εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα να προβώ σε κάποιες ε, συγκεκριμένες συστάσεις που θα φέρουν σε αντίθεση την κοινωνία των πολιτών με τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, Αντίθετα, θέλω να τονίσουμε τα κοινά συμφέροντα. Αλλά είναι βέβαιο ότι απαιτείται η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των παιδιών, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά στην επικράτεια της Ένωσης θα προστατεύονται. Και πράγματι, το να έχουμε διάφορες χώρες με διάφορους κώδικες διεντολογίες και, διάφο και διαφορετικούς κανόνες ε, περιπλέκει βέβαια τα πράγματα. Ενώ αν υπήρχε ε, μια, ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού και διαμόρφωσης των ε, κανόνων, αυτό πραγματικά θα μπορούσε να επιφέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Λίβενς. Νομίζω ότι το τελευταίο σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο περισσότερο υπάρχει κατακαιρματισμός του τοπίου, όσο περισσότερο επιβάλλονται διαφορετικές ε, υποχρεώσεις σε διάφορους παράγοντες και φορείς, τότε η, λύση που, προκρίνεται είναι συνήθως η απλούστερη, η ευκολότερη. Που στο, θέμα που συζητούμε είναι ότι απλώς οι εταιρείε απαγορεύουν την πρόσβαση ε, των παιδιών στα προϊόντα τους. Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο. Αν δείτε ε, τον, κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στόχος αυτού ήταν να προστατεύεται με ενιαίο τρόπο, με ομοιόμορφο τρόπο, ε, η προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Αυτό είναι δύσκολο βεβαίως καθήκον ε, και για τους αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όμως είναι και ένα περίπλοκο καθήκον και για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα και από μένα. Νομίζω ότι έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. σημειώσατε ότι βρισκόμαστε σε ένα, μια, ένα δύσκολο σημείο ως πολιτική. Αφενός θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, αφετέρου όμως δεν θέλουμε να πετάξουμε το παιδί μαζί με τα νερά και να παραβιάσουμε θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατακτήσουμε μια συνολική αντίληψη και κατανόηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και πράγματι έχουμε, έχουμε τα πράγματα είναι εύκολα. Όταν το, το περιεχόμενο είναι παράνομο, πρέπει να διαγράφεται τελεία. Πιο δύσκολο είναι όμως να ορίσει κανείς ποιο είναι το επιβλαβές περιεχόμενο. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να συνυπολογιστεί ότι και στη βάση πολιτιστικών ιδιομορφιών ε, τα διάφορα κράτη-μέλη αξιολογούν διαφορετικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα όρια της πορνογραφίας. Εδώ οι αντιλήψεις στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετικές. Και είναι πραγματικά δύσκολο να βρεθεί μία απάντηση. Για παράδειγμα, το βασικό ένστικτο που σήμερα πια θεωρείται κλασική ταινία στις ΙΠΑ ήταν ε, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, σχεδόν προκάλεσε σκάνδαλο. Όχι όμως λόγω των, ε, των σκηνών, των βίαιων, αλλά των ε, σεξουαλικά φορτισμένων σκηνών αυτής της ταινίας. Και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως υπάρχουν διαφορετικές διαφορετικέ αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Το να προσδιορίσουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι βλαβερό ως περιεχόμενο και το να καταλήξουμε σε μια πανευρωπαϊκή αξιολόγηση του τι τελικά είναι βλαβερό και τι όχι, αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλα αυτά βεβαίω συνδέονται και με το πώ θα διαμορφωθεί τελικά αυτός ο κώδικας διοντολογία, που βεβαίω θα πρέπει, θα πρέπει στη συνέχεια και να εφαρμόζεται. Αν όμω οι αξιολογήσει, οι αξιολογικές κρίσεις εκ των προτέρων είναι διαφορετικέ στα διάφορα κράτη-μέλη, βεβαίω καταλαβαίνετε ότι περιπλέκονται τα πράγματα. Κύριε Λίβινγκστον, ναι, πράγματι είναι μεγάλη πρόκληση αυτή. Η Ευρώπη βεβαίω δεν έχει κοινή αντίληψη ε, ως προς την ανατροφή των παιδιών και ποιες είναι οι κατάλληλες αξίες για τα παιδιά που πρέπει να, ε, να εμφυσίσουμε στα παιδιά. Ωστόσο, υπάρχει εμπειρία όσον αφορά την αξιολόγηση ε, του περιεχομένου. Υπάρχει και μια σχετική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εξετάζει ακριβώς αυτό στην εναρμόνιση των συστημάτων, όχι για να καταλήξουμε όλοι στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ώστε όλοι να έχουν κοινά εργαλεία, να υπάρχουν κοινέ ε, συζητήσεις και, και στη συνέχεια αφού θα τηρούνται κάποια ελάχιστα πρότυπα, κάποιες ελάχιστες προσδιαγραφές, να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη και τις, ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ε, τα πολιτιστικά και να καταλήγουν ε, στις ε, αποφάσεις τους. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε και κώδικα διδαντολογίας αλλά με μια ευελιξία. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι θετική. Αισιόδοξη είμαι. Βεβαίως θα απαιτηθεί πολιτική βούληση για να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως θα απαιτηθούν και μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή και την επιβολή αυτών των προδιαγραφών και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι και το κοινό θα κατανοεί πλήρω αυτέ τι προδιαγραφέ. Ε, Βεβαίω υπάρχουν και διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά ε, τον, τον πολιτισμό ή το επίπεδο των ψηφιακών ε, δεξιοτήτων. Ε, εδώ βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει ε, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Ωστόσο, από παντού ακούγεται πάντοτε ότι η παιδεία είναι, είναι η απάντηση. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακού αλφαβητισμού και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να τεθεί επικεφαλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να προσθέσω απλώς σχετικά με την αξιολόγηση του περιεχομένου. Είναι πολύ θετικό ότι στην πρόταση για, τις, για τη νέα οδηγία για τις ακουστικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται αυτό, το σύστημα δηλαδή περιγραφής του περιεχομένου. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το έργα νομίζω ότι θα είναι το φόρουμ όπου θα γίνει αυτό. Ένας χώρος δηλαδή όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν πώς ακριβώς θα χρησιμοποιούν αυτές τις περιγραφές του περιεχομένου. Αυτό από τη μία πλευρά. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι ότι αν επιβάλλουμε αυτά τα συστήματα περιγραφής περιεχομένου χωρίς συντονισμό, θα προκληθεί συντονισμός. Άρα χρειάζεται στρατηγική για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά βεβαίω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό, να υπάρχουν κοινοί κανόνε, γιατί το ίδιο περιεχόμενο που θα, θα μπορεί κανεί να, να το προσπελάσει από, διάφορες, ε, από διάφορα τεχνολογικά, τεχνολογικά μέσα. Άρα, θα πρέπει ε, να υπάρξει συντονισμός και συζήτηση με όλες τις φορές χάραξης πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλους τους εμπειρογνώμονες για αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι μας δώσατε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και τονίσατε ότι σημαντικό είναι γενικά, σημαντικότερο στοιχείο είναι γενικά ο αλφαβητισμός γύρω από τα μέσα επικοινωνίας όχι γιατί θα αποτελέσει την πανάκια ή τη μόνη λύση, αλλά επειδή αποτελεί δομικό στοιχείο προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους στο διαδίκτυο. Και βεβαίως αναδείξατε και τις ευκαιρίες, όχι μόνο τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που μας προσφέρουν αυτά τα μέσα επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την, παρουσίαση, για την παρουσία σας εδώ. Θα μας βοηθήσουν όλα αυτά που μας είπατε στο από εδώ και πέρα έργο μας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στην ε, εργασία σας από εδώ και πέρα. Και εμείς λοιπόν περνάμε τώρα στη συνάντηση των συντονιστών αλλά πριν από αυτό να σας, δώσω κάποιες, να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις επόμενη συνεδρίαση που προβλεπόταν να γίνει στις 5 Μαρτίου επειδή κάναμε τόση πολλή δουλειά τις δύο τελευταίες μέρες ακυρώνεται. Επομένως θα τα ξαναπούμε 19 Μαρτίου 3 με 6.30 το απόγευμα και 20 Μαρτίου ολόκληρη τη μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 6.30 το απόγευμα. Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσω βεβαίως όπως πάντα και τους ε, διερμηνείς και συνεχίζουμε μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα με την ε, συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.